Τη διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και ελπίζω ότι θα λάβουμε πλειοψηφία από αυτό το κοινοβούλιο στην ευρύνη ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μακάρθη. Ε, κλείνει η συζήτηση. Αύριο 11.30 θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία και προχωρούμε τώρα στην ε, ε έκθεση για δεύτερη ανάγνωση της κυρίας Γκρέσλε έρευνε που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατά πολέμηση τη Όλαφ. Η κυρία Γκράσινε, τέσσερα λεπτά. Είστε ταχύτερος από ό,τι φανταζόμουν. Ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάμε σε μια δύσκολη φάση σχετικά με τον κανονισμό για την Όλαφ ε, και τα εσωτερικά προβλήματα και λόγω ε, λαθών διοίκησης έχουμε προβλήματα και με την Επιτροπή Εποπτείας. Θα ήθελα να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τη δομή του αξιώματος που μας προβληματίζει, η δομή από την ίδρυσή του ε, δεν ταιριάζει στα δικαιικά συστήματα των κρατών μελών και γι' αυτό δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα που μέχρι τώρα ανεπαρκώς λύθηκαν και με τη μεταρρύθμιση, την αναμόρφωση. Ε, μέχρι τώρα κανονισμός της Όλαφ ε, όλα τα προσαρμόζει στον Γενικό Διευθυντή και όπως προβλέπει ο τωρινός κανονισμός είναι παντοδύναμος και πανταχού παρών. Από το 99 ίσχυε αυτό και παραμένει το καθεστώς. Σε μια επίπονη διαδικασία εμείς στο Κοινοβούλιο το 2008 ε, εισαγάγαμε ελέγχους και ισορροπίες, πιο δημοκρατικές δομές που υποστήριξε τότε και ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής και αυτά θα, θα προστάτευαν και τον ίδιο το Διευθυντή υπεξεργαστήκαμε ε, τις αποφάσεις του δικαστηρίου, ε, είδαμε τη ε, νομιμότητα των διαδικασιών και των ερευνών και αυτό διήρκεσε πολλά χρόνια. Η Όλαφ μέχρι τώρα δημιουργήσε θύματα δυστυχώς με τις μεθόδους της και ε, ε, στενοχωρούσε να, να αυξάνεται, να βλέπω να αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων. Ε, υπάρχει ως βάση ένα κείμενο της Κομισιόν που προέβλεπαν εξάρτητους ε, ελέγχους. Οι τροπολογίες μας αφορούσαν τους ελέγχους και τις ε, ε ισορροπίες που θα έπρεπε να τις διασφαλίσουμε. Ε, προέκυψε νέος ε, γενικός διευθυντής, ο οποίος ε, τις τροπολογίες που πρόβλεπαν τους ελέγχους και τις ισορροπίες τις απέρριψε. το ίδιο και ίσχυσε και για τις νέες διαδικασίες. Τώρα έχουμε μια δομή που περισσότερο από ποτέ στηρίζεται σε ένα μονοπρόσωπο και είναι όμοιρο στα χέρια του. Ε, αυτό το πρόσωπο δημιουργεί δυσκολίες και στην Επιτροπή Εποπτείας. Με την ευθύνη μου ως εισηγήτρια και επειδή γνωρίζω πολύ καλά το αξίωμα αυτό, ε, υπέβαλα κάποιες τροπολογίες για δεύτερη ανάγνωση. Ε, σκεφτείτε πολύ καλά πριν τις απορρίψετε γιατί μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τροπολογίες που στοχεύουν σε ένα πρόσωπο αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι εδώ υπάρχουν διαρθρωτικά λάθη στην δομή του αξιώματος και το κείμενο αναθεώρησης ενισχύει μάλλον αυτά τα διαρθρωτικά λάθη παρά τα αμβλήνη. Θέλω να σας καθησυχάσω. Η δεύτερη ανάγνωση μας δίνει τη δυνατότητα της συνδιαλλαγής. Μπορεί να τελειώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου έκανα 11 τριμερείς διαλόγους, 11 τριμερείς διαλόγους και στους 10 καθόμουν μόνη μου. Ο, Μπαρτ με βοήθησε. Ε, ε, δεν είχα πολύ βοήθεια. Ακόμα και όταν ζήτησα βοήθεια δεν με βοήθησε κανείς. Νομίζω ότι οι τροπολογίες είναι προς το συμφέρον του Συμβουλίου και γι' αυτό δεν θεωρώ ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι ε, εχέφρονες άνθρωποι στο Συμβούλιο και δεν νομίζω ότι ε, θα προχωρήσουμε σε περισσότερες από τρεις μήνες καθυστέρηση. Σημαντικό είναι ότι το κείμενο της αναμόρφωσης δεν λύνει τα προβλήματα, ενώ εγώ θα προτιμούσα να λυθούν κάποια ή ένα τουλάχιστον το θέμα της νομιμότητας των διαδικασιών και η πρόσβαση της Επιτροπής Εποπτείας. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να λυθούν τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι το κείμενο ε, είναι καλύτερο από την αναμόρφωση που είχε πραγματοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε και τώρα ο Επίτροπος Σέμετα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Σήμερα συζητάτε το κείμενο για την αναθεώρηση της νομικής βάσης όσον αφορά την Όλαφ μετά από πολλές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο που προχώρησαν 7 ολόκληρα χρόνια. Και το έργο συμβιβασμού είναι αυτό που έχετε μπροστά σας, με το οποίο συμφώνησαν στο τριμερή διάλογο το 2012 τα τρία θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λέει ότι είναι τέλειο το τελικό κείμενο, είναι όμως ένα πολύ καλό αποτέλεσμα το οποίο πετύχαμε μετά από έντονες διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων των πλευρών. Μην ξεχνάμε ότι ο συμβασμός αυτός θα βελτιώσει το έργο της Όλαφ. Οι βελτιώσεις αυτές είναι ουσιαστικές ιδιαίτερα για τα άτομα που τελούν υποδικητική έρευνα στην Όλαφ. Μέσω του νέου κανονισμού θα υποφελούνται από ενισχυμένες διαδικασίες προστασίας. Η νομοθεσία επίση διασφαλίζει διάφορου τρόπου με του οποίου μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η Όλαφ και να προστατεύει έτσι τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι πολύ σημαντικό τη σήμερα ημέρα για ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι αναγκαίο να εγκριθεί το κείμενο αυτό ως έχει. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν αντιλαμβανόμαστε και εμείς τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει όλους αυτούς τους μήνες πολλοί από εσά αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει περίοδο, περιθώριο βελτίωσης του έργου της Όλαφ και πέρα από την έκθεση αυτή. Παρ' όλα αυτά είμαστε πεπισμένοι ότι ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι βήμα-βήμα. Και ως πρώτο βήμα πρέπει να διασφαλίσουμε αυτό που έχουμε πετύχει στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε την αναθεώρηση του κανονισμού για την Όλαφ άνευ κάτι το οποίο θα επιτρέψει στη ρύθμιση αυτή να αρχίσει να ισχύει τους επόμενους μήνες και έτσι να έχουμε πολύ γρήγορα βελτιώσεις. Δεύτερο βήμα. Να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε το νομικό πλαίσιο της Όλαφ ακόμα περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπόψη της δύο στοιχεία. Μετά από την πρόταση που υπάρχει όσον αφορά την Υπηρεσία Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Το πρώτο βήμα θα ήταν να υπάρξει ένας ανεξάρτητος επόπτης. Το άτομο αυτό θα μπορούσε να ελέγχει κατά πόσο τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων που τελούν υποδικητική έρευνα. Και δεύτερον, να δούμε τα ερευνητικά μέτρα. Κατά πόσο δηλαδή γίνονται έρευνες σε γραφεία, σε έγγραφα, η υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα χρειάζεται δική για να προβεί σε τέτοια μέτρα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τα ερευνητικά μέτρα της Όλαφ θα πρέπει επίσης να ε, υποβάλλονται σε μια ειδική διαδικασία. Θέλουμε να επικεντρωθούμε επίσης στην Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ, η οποία έχει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι απαραίτητα το κατάλληλο όργανο για να αναλάβει τα δύο αυτά νέα μέτρα στα οποία αναφέρθηκα και ποτέ δεν ήταν αυτός ο στόχος της Επιτροπής αυτής, να κάνει δηλαδή προσωπικές έρευνες. Είναι επιπλέον από τις αρμοδιότητές τους και έπειτα δεν υπάρχει καμία νομική ευθύνη ώστε να μπορούν τα μέλη της Όλαφ να προβούν σε τέτοιες έρευνες. Εμείς πιστεύουμε ότι η συνεργασία με την Όλαφ και την Εποπτική Επιτροπή πρέπει να βασίζεται σε σαφείς και από τις δύο πλευρές ε, συμφωνισμένα μέτρα και αρχές. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία με αντικειμενικότητα και ο κοινό μα στόχο να είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα λειτουργεί αποτελεσματικά, ότι προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο που έχουν θέσει οι ίδιοι νομοθέτε. Και συγχρόνω πρέπει να σκεφτούμε και νέε εναλλακτικέ λύσει όπω αυτέ που σα περιέγραψα πριν από λίγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προωθήσει το έργο αυτό ω προτεραιότητα σε συνεργασία πάντα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ουσιαστική πρόοδο που επετέφθη στι συζητήσει που έγιναν τα τελευταία αυτά χρόνια για να βελτιωθεί το πλαίσιο εργασία τη Όλαφ, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για παράδειγμα, είναι κάτι που πρέπει να γίνει νόμος χωρί άλλη καθυστέρηση. Ελπίζω, συνεπώ ότι θα στηρίξετε το κείμενο το οποίο ενέκρινα τα τρία θεσμικά όργανα και θα συμφωνήσετε να προχωρήσουμε στην επικοδομητική μα συνεργασία για να λυθούν τα εκκρεμούντα ζητήματα με τον καταλληλότερο τρόπο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε Σέμετα και τώρα οι αγορητές εξ των ομάδων ο συνάδελφος Ντόιτς για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα συνοψίσω σε τρία σημεία αυτά που θέλω. Καταρχήν να σας πω ότι η μεταρρύθμιση, η αναμόρφωση της Όλαφ, το σχετικό κείμενο και η συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο τώρα λαμβάνουν χώρα κάτω από διαφορετικά δεδομένα. Μετά την απαραίτηση του Μαλτέζου Επιτρόπου και μετά τα διαδικαστικά προβλήματα που προέκυψαν. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για Dali Gate, αλλά μάλλον για Olaf Gate. Η πληροφο... Πάνω στη βάση των πληροφοριών φάνηκε ότι, γενικός... ότι ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ ε, διέπραξε σημαντικές παρατυπίες που αν επρόκειτο για άλλον αξιώμα του από κάποιο κράτος μέλος θα συνεπαγόταν απευθείας ε, παρέτηση ή απόλυση. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, δεν ε, μπορώ να συμφωνήσω με τον Επίτροπο Σέμετα. Συνήθως λέμε στην Ουγγαρία ότι δεν μπορούμε ένα χάσμα να το περάσουμε ε, με ε, ε, κομματάκια, λεπτά κομματάκια ξύλο γιατί θα πέσουμε στην Άβυσσο. νομίζω ότι θα έπρεπε να έχω τρία λεπτά γιατί έτσι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ. Ωραία, συνεχίστε λοιπόν. ευχαριστώ πολύ. Η εφαρμογή της ε, αναμόρφωσης της όλα δεν μπορεί να γίνει σταδιακά. Γι' αυτό υποστηρίζω σε μεγάλο βαθμό και την έκθεση της κυρίας ε, Γκρέσλε και τις τροπολογίες. Σε τελευταία ανάλυση, κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι το εξής. Αν ε, αύριο στην Ολομέλεια δώσουμε μια απάντηση που δεν δώσει νέα κίνητρα για την αναμόρφωση αυτή, τότε θα... Ε, αυτό το, αυτή η υπηρεσία που δημιουργήθηκε το 1999 και που με τις δραστηριότητες του ε, ε, έκανε πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή ε, βοήθησε τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν δεν δώσουμε λοιπόν αύριο με την ψηφοφορία μας νέα κίνητρα για την αναμόρφωση, η Όλαφ δεν θα είναι μέρος της λύσης αλλά του προβλήματος. Ελπίζω λοιπόν ότι αύριο θα εγκρίνει την έκθεση αυτή το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάιερ δύο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Σέμετα, αγαπητοί συνάδελφοι. Αύριο θα αποφασίσουμε αν ε, συμφωνούμε με τον τριμερή διάλογο για την Όλαφ ή όχι. Και εγώ πρέπει να πω ότι είμαι. Κάναμε πρόοδο εκεί που χρειάζεται, ε, ορισμένες βασικές έννοιες ε, ξεκαθαρίστηκαν, η πρόσβαση στα δεδομένα από την Όλαφ είναι ρυθμισμένη. Υπάρχουν διαδικαστικές, διαδικαστικά ε, πλεονεκτήματα και προστασία. Υπάρχουν συγκεκριμένες ε, διατάξεις για τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ο οποίος παρακολουθεί και εξασφαλίζει την νομιμότητα και ε, καταρτίζει ένα πλαίσιο για τις έρευνες της Όλαφ. Όλα αυτά είναι σημαντικά, είναι πρόοδος και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, την κυρία Γκρέσλε και τον σκιώδη εισηγητή, τον κύριο Μπαλτσίτης. Ε, υπάρχουν αρκετές τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι είναι αθέμητες ή αντικειμενικά λανθασμένες. Μεταξύ αυτών ε, έχουμε και τροπολογίες από την ομάδα μου αλλά δεν μπορούμε να ε, κλείσουμε τα μάτια στους κινδύνους από τις περαιτέρω διαδικασίες. Η Κομισιόν μετά από 7 χρόνια ε, θέλει να θέσει σε εφαρμογή την ε, νομοθεσία. Η, η Ιρλανδική Προεδρία δεν μας ενημέρωσε σχετικά με την απροθυμία να ανοίξει το θέμα αυτό. Ε, στις 2 Οκτωβρίου του 2012 μας είχαν κοινοποιήσει ότι αν δεν γίνει η διαπραγμάτευση αποδεκτή τότε θα αποσύρουμε την πρόταση και αυτό είναι μια οπισθοχώρηση σε σχέση με τις βελτιώσεις που είχαμε τόσο δύσκολα επιφέρει. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ε, ε, τις πρόοδους ε, ορισμένες τροπολογίες ε, του ΕΛΚ πρέπει να τις ε, απορρίψουμε διότι πιστεύουμε ότι δημιουργούν κινδύνους για την όλα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μούλτερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κρίμα που και μετά τις τελευταίες παρατηρήσεις του κ. Γκέι δεν έχουμε εδώ και άλλους αξιωματούχους. Συγχαρητήρια στην Ingeborg Gressler πάντως όπως συνήθως και αυτή τη φορά έφερε σε πέρας αυτό που ανέλαβε με πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, έχουν συμβεί και διάφορα με τον Επίτροπο Νταλή. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι οι τροπολογίες που προτείνει δεν είναι κακές. Το μόνο το οποίο εμένα με απασχολεί είναι πώς θα εξετάσει το Συμβούλιο, τι θα κάνει το Συμβούλιο στη συνέχεια με αυτά. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Η σχέση ανάμεσα στην Επιτροπή Εποπτείας και την ίδια την Όλαφ. Και γι' αυτό θα ήθελα να έχω την άποψη του Επιτρόπου. Μήπως θα έπρεπε σύντομα να, υπάρξουν, να υπάρξει κάποιος ορισμός κάποιου ανεξάρτητου, ο οποίος θα φροντίσει για την ε, εποπτεία και θα προστατεύσει έτσι την Όλαφ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάις έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αύριο έχουμε δύο επιλογές, συνάδελφοι. Ή που εγκρίνουμε τις τροπολογίες της κυρίας Γκρέσλερ, Βοβέ, Γιόγκε κλπ. Ή απορρίπτουμε το κείμενο. Και τι λένε οι τροπολογίες, προσπαθούν να μας διδάξουν από αυτά που είχαμε μέχρι τώρα διαπιστώσει. Τα... Το παίρνουμε το μάθημα από τις ε, δραστηριότητες της εποπτείας στην Όλαφ και το αναφέρονται στο παράρτημα 3. Δεν μπορούμε να νομοθετούμε από το τίποτα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αντίφαση εδώ ανάμεσα τον επικεφαλής της Όλαφ και της Επιτροπής Εποπτείας. Άρα πρέπει να δούμε κατά πόσο ακολουθούνται οι διαδικασίες και πώς θα το πετύχουμε αυτό και ποιος είναι υπεύθυνο. Αύριο λοιπόν συνάδελφοι έχουμε δύο επιλογές. Ή που εγκρίνουμε τις τροπολογίες και τότε είμαστε σε ισχυρή θέση απέναντι στο Συμβούλιο ή λέμε ας πάμε στη διαδικασία συνδιαλλαγής χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό όμως που θέλουμε. Οπότε δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν μια ομάδα δηλών. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε στο Συμβούλιο κάντε αυτό που εμείς έχουμε αποφασίσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγκρίνετε τις τροπολογίες τις δικές μου του κ. Ποβέ, του κ. Ντογιόνγκη και τις της κυρίας Κρέσλη και ας δείξουμε ως Κοινοβούλιο ότι έχουμε την πυγμή να επιβάλλουμε τη θέλησή μας. Ευχαριστώ. πολύ. Ο κύριος Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Στασί είπε όλα ήθελα να πω και εγώ. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη υποπτία της Όλαφ και τα λοιπά. Αλλά ας μιλήσουμε εδώ πιο συγκεκριμένα. Έχουμε κάποιες τροπολογίες που μπορεί να θεωρηθούν ως εργαλεία για την Όλαφ να βελτιωθεί, να είναι πιο αποτελεσματική. Αλλά επίσης να καταστεί και πιο εύκολος ο έλεγχος. Κατά την άποψή μου, το να δώσουμε περισσότερα εργαλεία στην ε, Επιτροπή Εποπτείας ε, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν ε, υιοθετηθούν αυτές οι τροπολογίες, εμείς θα τις υποστηρίξουμε και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τις υποστηρίξει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσαρνέτσκι. Ο κύριος Ντεγιόγκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα τους συναδέρφους Χρέσλερ και Στάες. Η κατάσταση στην Όλαφ είναι σοβαρή. Πρώτον, υπάρχει λύση όσον αφορά τη διαμάχη με την Επιτροπή Εποπτείας. Όπως λέει και ο κύριος Μέλντερ, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί τελικά αυτή η Επιτροπή και να βελτιωθεί η λειτουργία της ακόμα περισσότερο. Έπειτα, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται απομακρύνονται πολύ από τα κράτη-μέλη, έτσι είπε ο Επίτροπος. Τα κράτη-μέλη το αντιλαμβάνονται αυτό. Μήπως πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη εξωτερική έρευνα. Η πίεση της Επιτροπής πάνω στην Όλαφ, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά, έχω μιλήσει με την κυρία Κρέσλερ. Πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμα. Για μένα απλώς τώρα αναβάλουμε ακόμα περισσότερο τη δράση μας, ενώ θα έπρεπε να δράσουμε άμεσα. Ευχαριστώ. Κύριος Χάρτονγκ, ένα λεπτό. Συνέδερφο Γκρέσλερ, πολύ καλά κάνετε και βάζετε στο μικροσκόπιο τις δραστηριότητες της Όλαφ. Δεν λειτουργεί καλά. Είναι σοβαρό όμως ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Αυτός είναι και ο ρόλος της Όλαφ, άρα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά όλα αυτά. Από ίδια εμπειρία, ξέρω πριν από χρόνια για μια περίπτωση διαφθοράς, η Όλαφ έκανε την έρευνα και τελικά δεν βρήκε τίποτα, ούτε καν ε, δείγματα. Πρόεδρε, είναι πολύ σοβαρό όλα αυτά. Υπάρχουν ένα σωρό υποθέσεις στο γραφείο της Όλαφ και δεν πιστεύω ότι ποτέ θα διεκπαιρεθούν. Σήμερα λοιπόν δεν πρέπει να μιλάμε για μια καλύτερη Όλαφ, αλλά μήπως να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Πάρα πολλά χρήματα σπαταλώνται και δυστυχώς η διαφθορά είναι πάντα παρούσα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τους ομιλητές για τις πολιτικές ομάδες ε, οι υπόλοιποι ομιλητές τώρα. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ο ελευθερημένος κανονισμός εδώ σε σχέση με την Όλαφ ε, θέλει να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στην Όλαφ να είναι πιο αποτελεσματική για την καταπολέμηση της απάτης και δυστυχώς ε, ε, αυτό μπλοκάρεται κυρίως ε, στην περίπτωση των ερευνών κατά του κυρίου Ντάλι που δεν ήταν και τόσο ευτυχής ε, δυστυχώς ε, και φυσικά το πώς η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ και ο κύριος Κέστλερ υλοποίησε τις έρευνες. Υπήρξαν κάποιοι εριστεχνισμοί όμως πρέπει να ε, προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, είναι απαραίτητες και μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την ενδυνάμωση της Όλαφ. Επίσης να προστατεύσουμε όσους κρούν το κονδύνο του κινδύνου, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Όλαφ και των κρατών μελών, μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Όλαφ και ενδυνάμωση της Επιτροπής Εποπτείας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Και τώρα ο κύριος Μπαλτσίτης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε για την εξαιρετική δουλειά της ε, και ε, το στόχο της να ενδυναμωθεί η ΟΛΑΦ, ε, ένας οργανισμός που είναι απαραίτητος για την καταπολέμηση της απάτης και την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δυστυχώς ε, βλέπουμε ότι ε, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των απατών πρέπει να ενδυναμώσουμε την ΟΛΑΦ. Η έκθεση θέλει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της Όλαφ και λυπάμαι που σήμερα στις συζητήσεις μας επικεντρωνόμαστε σε διαφωνίες μεταξύ της Όλαφ και της Επιτροπής Εποπτείας και της ανικανότητάς τους να κατανείμουν τις αρμοδιότητές τους παρά στην ε, μεταρρύθμιση της Όλαφ που αποτελεί αποτέλεσμα 7 χρόνων σκληρής δουλειάς στην εργάζονται περίπου 500 άνθρωποι και δεν νομίζω ότι ε, θα πρέπει η δουλειά τους να παρεμποδίζεται ε, λόγω διαθεσμικών διαφωνιών. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία της Όλαφ και των υπόλοιπων φορέων και θα πρέπει να προστατεύουμε τα δικονομικά δικαιώματα των ανθρώπων ε, που είναι υπό έρευνα. Μπορεί το κείμενο που έχει συμφωνηθεί να μην είναι ιδανικό για κανένα μέρος, αλλά οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα ποιότητα των ερευνών τη ε, Όλαφ. Η τέλεια μεταρρυθμίση δεν υπάρχει, όμως η μεταρρυθμίση τη Όλαφ θα είναι το πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των δραστηριοτήτων της ε, και την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της. Ως κοιόδης εισηγητής έχω κατά νου τον ρεαλισμό και προτείνω να υιοθετήσουμε το κείμενο έτσι όπω έχει συμφωνηθεί με το Συμβούλιο, δηλαδή χωρί τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Μπαλτσίτη. Ε, Τέχεστε ερώτηση από τον κύριο Στάς. Παρακαλώ, συνάδελφε Στάση. Συνάδελφε Μπαλσίτης, είσαστε ένας σοφός άνθρωπος, ένας πολύ καλός συνάδελφος, αλλά δεν καταλαβαίνω τη στάση της ομάδας σας. Έχουμε μια διαδικασία να νομοθετούμε σε τρία στάδια με τη δεύτερη ανάγνωση μετά πάμε σε συνδιαλλαγή. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές έχω συμμετάσχει κι εγώ. Και όπως λέει και η κυρία Γκρέσλερ, η συγκήτρια σε τρεις μήνες θα έχει ολοκληρωθεί. Αν τώρα εγκρίνουμε τη δεύτερη ανάγνωση, τότε θα αργήσει πάρα πολύ η εφαρμογή. Διακόπτει το μικρόφωνο ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Στάς. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, γι' αυτό παρακαλώ συντομεύετε. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα επί ώρες. Η Κομισιόν εξήγησε πολύ καλά τη διαδικασία ίσως να μην έχουμε τρεις μήνες. Αυτή η μεταρρύθμιση μπορεί να αναβληθεί για δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, εκτός και αν κατορθώσουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία τώρα. Αυτές τις πληροφορίες έχω εγώ και γι' αυτό ανέφερα τη θέση του κ. Γκάι του συντονιστή μας. Ο Επίτροπος υποσχέθηκε γραπτός ότι αμέσως ε, μετά την έγκριση της συμφωνίας αυτής θα περάσει στο επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε κύριο Στόιρε. Ένα λεπτό. Ε, πραγματικά είμαστε σαν ε, σε τραγωδία του Σέξπιρ μπροστά σε κρίσιμη καμπή. Το θέμα είναι αν θα έχουμε λειτουργική ε, επιτροπή εποπτείας ή όχι. Από πέρσι τον Οκτώβριο Είχα συμφωνήσει με την εισηγήτρια έξι χρόνια το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, έδωσαν μάχη για μια συμβιβαστική λύση. Τον περασμένο μήνα ε, η ε, τα θεσμικά όργανα ε, παρουσίασαν ε, όλες τις δυσκολίες της Όλαφ. Δεν μπορώ να φανταστώ να μην έχει Επιτροπή Εποπτείας. Άκουσα ότι υπήρχαν συνεννοήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κυρίου Μπαρόζο και των Ευρωβουλευτών. Είμαστε επιτέλους έτοιμοι να ε, ζητήσουμε την ανεξαρτησία της Επιτροπής Εποπτείας μπορείτε να μιλήσετε στο Συμβούλιο όπως εδώ σε εμά. Δεν μπορεί να υπάρξει αναμόρφωση της όλα χωρίς να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής ε, Εποπτείας. Ευχαριστώ πολύ ε, και για την αναφορά στον Σέξπιρ. μπορεί να υπάρχει τρέλα, αλλά υπάρχει μέθοδος αυτήν. Η συνάδελφος Ανδρέασεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν κάποιος χρειαζόταν αποδείξεις για το πόσο αναποτελεσματική είναι η θεσμή της Ένωσης, ε, ειδού τα 7 χρόνια που χρειάστηκαν για το ρυθμιστικό, κανονιστικό πλαίσιο της, για την αναμόρφωση της Όλαφ. Ακόμα και όταν έχει βρεθεί συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, υπάρχει ανάγκη και για άλλες τροπολογίες. Το πιο σημαντικό όμως είναι η ανεξαρτησία της Όλαφ, αυτό το πλαίσιο δεν την εξασφαλίζει σωστά. Τη Όλαφ ε, στόχο έχει να, καταπο... να, να... συμβάλλει στην αποφυγή ε, απατών. Ε, εξορισμού λοιπόν πρέπει να είναι ανεξάρτητη Όλαφ από τους ε, ε, φορείς που χειρίζονται κονδύλια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο επίσης. Η Όλαφ πρέπει να ε, αναφέρεται χωρίς ενδιάμεσους άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες που χρηματοδοτούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό και ο κανονισμός της δεν πρέπει να υπόκειται. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε συνάδελφε Ανδρέασεν και πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Φίγκετ ζητεί μόνο το λόγο. Θέλω να πιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημαντικό θέμα το οποίο δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα στη συζήτησή μας. Οι δραστηριότητες της Όλαφ έχουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για τους πολίτες της Ευρώπης, οι οποίοι θα διαφερθούν ακόμα περισσότερο το 2014, το έτος δηλαδή των ευρωπαϊκών εκλογών. Γι' αυτό πιστεύω ότι η εκστρατεία πληροφόρησης όσον αφορά την Όλαφ θα έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να έχουμε κοινέ προδιαγραφές για το τι πληροφορίες και πώς οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιοποιούνται γιατί φοβάμαι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο που έχει η ενημέρωση αυτή. Και συχνά πρώτα πηγαίνει στον τύπο και μετά αποφασίζουμε εμείς τι θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε και πώς. Ευχαριστώ κύριε Σέμκε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο κυρία Σέμετα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα κύριοι βουλευτές. Είναι σαφές ότι και αυτός ο οίκος και η Κομισιόν έχουν τον ίδιο στόχο σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της Όλαφ και δύο σκοπεύουμε στο να βελτιώσουμε το νομικό πλαίσιο τη Όλαφ για να υπάρξει πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πραγματική παρακολουθήση από τι εθνικέ αρχέ και πιο αποτελεσματική εργασία του γραφείου και συστημική παρακολουθήση από την Επιτροπή Εποπτείας. Για να απαντήσω λοιπόν στον κύριο Τουιερνέ, είμαι υπέρ του να έχουμε ισχυρή Επιτροπή Εποπτείας. Παρ' αυτά, όπω ε, ήδη είπα στην εισαγωγή μου, είμαι πεπισμένο ότι μια προσέγγιση σε δύο βήματα είναι κατάλληλη και μάλιστα απαραίτητη για το φάκελο αυτό. Ως πρώτο βήμα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, σημαντική βελτίωση του νομικού πλαισίου της Όλαφ που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και για τις οποίες η δική σας συγγήτρια εργάστηκε πολύ σκληρά. Δεύτερο βήμα, η Κομισιόν δεσμεύεται να βρει τρόπους να βελτιώσει το νομικό πλαίσιο της Όλαφ ακόμη περισσότερο μόλις τεθεί ισχύ ο κανονισμό, Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να εμπνέεται από την πρόταση για την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα που θα θετήσει πρόσφατα η Κομισιόν ε, θα συμπεριλαμβάνει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ε, διοργανικής ανταλλαγής απόψεων. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να υποστηρίξει την προσέγγιση αυτή που είναι προς το συμφέρον και των ενδιαφέρον ατόμων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και νομίζω ότι διαφορετικά θα βιώσουμε τον κίνδυνο αντί να έχουμε άμεση υιοθέτηση του κανονισμού και σημαντική βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου της ΟΛΑΦ. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε επί της μεταρρύθμισης ε, και μάλιστα τέτοιες συζητήσεις μπορούν να διαρκέσουν 10-12 χρόνια. Αυτό είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε έμετα και στο τέλος της συζήτησης η εισηγήτρια κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις. Θα ήθελα να πω το εξής. Όταν ψηφίσουμε τις τροπολογίες έχει τρεις μήνες χρόνο να τις εξετάσει το Συμβούλιο. Αν συμφωνεί εντάξει, αν δεν συμφωνήσει θα γίνει νέα διαδικασία συνδιαλλαγής. Θα καθίσουμε όλοι μαζί να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Και θα μπορέσουμε σιγά σιγά και με δυσκολίες να πείσουμε το Συμβούλιο. Αυτό υποθέτω. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο Γκίνσπερκ από τη Δανέζικη Προεδρία και τον κύριο Κρατσίνσκι από την Πολωνική Προεδρία. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τόσο πολύ το Συμβούλιο και εκείνο ενδιαφέρεται να βελτιωθεί η καταπολέμηση της απάτης ε, παρόλο που είναι δύσκολο να το δείξει αυτό. Ε, ε, εμείς πραγματικά έχουμε την ίδια κατάσταση όπως πριν από την ψηφοφορία το 2008. Είναι λίγο ε, κομικό αυτό. Ε, ακούγαμε από την Κομισιόν τότε ότι ήταν απίθανο αυτό που είχα υποβάλει ως πρόταση η, η Κομισιόν επί δυόμιση χρόνια είχε παγώσει όλο το φάκελο και δεν το επεξεργάστηκε καθόλου θεωρούσε ότι ήταν αδύνατον αυτό και τώρα ε, μπορέσαμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Καλό είναι τα προβλήματα που βλέπουμε εδώ και δύο χρόνια και τα βλέπουμε να παρουσιάζονται ξανά και ξανά. Έχουμε μια ευκαιρία να τα λύσουμε. Γι' αυτό παρακαλώ ας το δοκιμάσουμε, ας αποπειραθούμε δεν θα ε, εξαφανιστούν στο γάλαθο των σκουπιδιών όλα αυτά. Και μάλιστα καλό είναι να συμμετάσχουν στη συζήτηση και οι συνάδελφοι που ήταν και στις ε, προηγούμενες διαδικασίες ε, συνδιαλλαγής. Κύριε Σεμέτα, για την προσέγγιση των δύο σταδίων βημάτων, το 2006 η Κομισιόν είχε προτείνει ανεξάρτητο ελεγκτή το 2011 την αποσύρατε την πρόταση. Το 2014 θέλετε να την επανυποβάλλετε. Μα η υπόθεση αυτή είναι σοβαρή. Ήρθε τώρα η ώρα να ε, λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Αύριο στις 11.30 θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Τώρα, κοινή συζήτηση για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έκθεση του κυρίου Βόν